δικαιώματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θέλω να εκφράσω την θλίψη όλων μας για το θάνατο ενός αγαπητού συναδέλφου, του Μιγγέλ Σακαντούρα Πόρτας, ο οποίος στις 24 ε, Απριλίου σε ηλικία μόνο 53 ετών απέθανε. Ο συνάδελφος Πόρτας ήταν οικονομολόγος. Στη συνέχεια εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Ένα λειτουργήμα που ίσκησε ως δημοσιογράφος και το οποίο το έκανε με μεγάλη προσήλωση και με μεγάλο πάθος όπως γνωρίζουμε όλοι. Ο Μιγγέλ το 2004 για πρώτη φορά εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. σαν 15χρονος. Ο Μιγγέλ είχε συλληφθεί από την αστυνομία του Σαλαζάρ λόγω της συμμετοχής του σε μια φοιτητική διαδήλωση στο, στη Λισαβόνα. Έλαβε μέρος στην επανάσταση των Γαριφάλων που οδήγησε στην κατάρρευση της δικτατορίας στην Πορτογαλία. Όλη του η ζωή ήταν ένας παθιασμένος αγώνας ως αριστερού ακτιβιστή και ενός ένθερμου υπέρμαχου της δημοκρατίας. Γνώρισα τον Μιγγέλ Πόρτα σαν πεπισμένο Ευρωπαίο, ο οποίος αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν, όπως και άλλοι, στο ίδιο μήκος κύματος, δεν είχαμε τις ίδιες πεπιθήσεις, όλοι μας έχουμε αναγνωρίσει την επικοδομητική, την θετική, την ανθρώπινη του προσέγγιση σε θέματα που ήταν επίμαχα σε συζητήσεις που είχαν πολλές αντιθέσεις. Τον γνώρισα και τον έχω ζήσει σαν ένα συνάδελφο ο οποίος ήταν πάντα δίκαιος και σωστός και ο οποίος δεν υπεκρύφτηκε ποτέ πίσω από διαδικαστικά θέματα, προσπάθησε πάντα να εξασφαλίσει δημοκρατικές πλειοψηφίες και ήταν πάντα έτοιμος να δεχθεί την ήττα του όταν δεν το επιτύχαινε. Αλλά ήταν πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος τήρησε το λόγο του για όλους μας είναι ένα άτομο το οποίο δεν θα το λησμονήσουμε. Ο Μιγγέλ ήταν ένας από τους συναδέλφους μας, ο οποίος μπορούσε να αυτοσατηρίζεται ακόμα και να αναγνωρίζει τα δικά του λάθη χωρίς πρόβλημα. Οι σκέψεις μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές βρίσκονται με την οικογένειά του και τους φίλους τους και αύριο θα υπάρξει και μια τελετή στην μνήμη του Μιγέλ Πόρτα στο Κοινοβούλιο, στην οποία είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Έχουμε χάσει πράγματι ένα εξέχοντα ε, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μια ύπουλη ασθένεια ενάντια στην οποία αγωνίστηκε θαραλέα αλλά τελικά έχασε τη ζωή του και έχουμε χάσει ένα πάρα πολύ αξιόλογο συνάδελφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής για ένα λεπτό Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.